Θα ήθελα να σε επιπλέον ότι ε, δήλωσα αποδεκτή την πρόταση πράξης της Ένωσης που τροποποιεί την ε, οδηγία για ένα κοινό πρόγραμμα ε, σύστημα μάλλον προστιθέμενης αξίας που επευλήθη από τον κύριο Σούλικ και αυτό λόγω των οικονομικών και νομισματικών